Ε, καλησπέρα σα, συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η σύνεδρος που διακόπη στις 16 του μηνό. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η Ολομέλεια. Καθίστε παρακαλώ και διακόψτε τις συνομιλίες. Σας ενημερώνω τα συνοπτικά πρακτικά της 16ης Νοεμβρίου είναι διαθέσιμα.